Ε, Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Μετά από τη μισάωρη διακοπή, ζητώ από όλους να καθίσουν παρακαλώ. Az képviselő képviselőcsoportnak volt egy kép... Η πολιτική ομάδα EFTD κατέθεσε ένα αίτημα. Διαδικαστικό, για διαδικαστικό ζητάτε το λόγο. Παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο. Κοιτάξτε, δεν με πειράζει αν ε, μου είπα να το βουλώσω όπως μου είπε ο αξιότιμος ε, κύριος του